Bien. Buena, buenos días a todos. Καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Σε σχέση με την πρώτη έκδοση της ημερήσιας διάταξης δεν είναι κάποια τροποποίηση γιατί υπήρξε αναγγελία. Σύμφωνα με το σημείο 9, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αλία με το Μαρόκο, και όπως ε, είχαμε και στην ίδια ημερήσια διάταξη, αν δεν υπήρχαν τα έγγραφα, έγγραφα διαθέσιμα δεν θα, τα, δεν θα το εξετάζαμε, δεν είχαμε τα έγγραφα λοιπόν διαθέσιμα και αναβάλλεται αυτό το θέμα 9 για τη συνεδρίασή μας του Οκτωβρίου. Καταρχήν δεν υπάρχει καμιά άλλη ε, τροποποίηση της ημερησία διάταξης ή άλλη προσαρμογή καθότι γνωρίζουμε. Λοιπόν, μια και συμβαίνει αυτό, περνάμε στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχουμε αυτή τη στιγμή και υπό τα διάφορα αν χρειάζεται κάτι μπορούμε να κάνουμε κάποια παρατήρηση, κάποια αναγγελία. Και περνάμε ήδη, αν συμφωνείτε, στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι ετοιμάστε τις κάρτες σας για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ετοιμαστείτε είναι οι γνώσει ε, για τον θαλάσσιο, το θαλάσσιο περιβάλλον, για τη θάλασσα, βελτίωση της χαρτογράφησης ε, του βυθού για αλληλευτικού σκοπούς για την αηφορία, έκθεση της κυρίας Πατράου. Υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποιο θέμα πριν ξεκινήσουμε με την ψήφιση. Αν όχι, ξεκινάμε άμεσα με την ψήφιση, την ψηφοφορία. Λοιπόν, συμβιβασμό υπαριθμών 1. Ξεκινάμε έτσι. συμβιβασμό 1 με τα χέρια ψηλά να πάμε ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε εγκρίθηκε λοιπόν συμβιβασμός 2 παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο Πάντα κανονικά σε αυτή την κοινοβουλευτική επιτροπή, κυρία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Εν πάση περιπτώσει συμφωνούμε όλοι γι' αυτό. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε πάντα. Πάμε πιο γρήγορα, εν πάση περιπτώσει, και δεν μετράμε, δεν καταμετρούμε ψήφου και χέρια κτλ. Αυτό κάνουμε. Συμβασμό 2. Ψηφίζουμε. Άρχεται. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίφθηκε η 11. 12 άρχεται. Τι είπατε εσείς. Εντάξει, 12 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 4. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 19. 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 5. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 6 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούστηκε. Εντάξει, το αποτέλεσμα λέτε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Θα το τακτοποιήσουμε αυτό, θα γνωστοποιηθεί Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 27. Πιο αργά να πηγαίνω, έτσι. Εντάξει, με βραδύτερο ρυθμό. Ωραία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 28. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Τροπολογία 29 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 30 άρχεται. η σοσιαλιστική ομάδα έχει έναν παραπάνω που συμμετέχει στην ψηφοφορία. Η σοσιαλιστική ομάδα έχει έναν παραπάνω στις ψήφους που καταμετρούμε. Τροπολογία 3, 30 εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 9. Άρχεται. Πέρας. Ένα σοσιαλιστής παραπάνω πάλι. Λοιπόν, θα επαναλάβουμε. Ξεκινάμε πάλι με το συμβασμό 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 10. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Και τώρα θα ψηφίσουμε το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ και μία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Πατράουν Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας. Σημείο 5. Προς μια σφαιρική ολοκληρωμένη αλευτική στρατηγική της ΕΕ στην περιοχή του Ατλαντικού. Ξεκινάμε με την ψηφοφορία. Τροπολογία υπαριθμών 23. Ναι. Ναι, εσείς. Έχουμε ένα συμβιβασμό 2. Θα λέγα δεν είναι πραγματικά συμβιβασμός. Έχουμε πρόβλημα με την ομάδα μου. Θα ψηφίσουμε επ' αυτού ή όχι. Τι θα κάνουμε για το συμβιβασμό 2. Διότι αναφέρομαι και εγώ εκεί. Λοιπόν, πρόεδρος, θα το δούμε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε όπως γίνεται με τους συμβιβασμούς Καμιά φορά κάποιοι δεν συμφωνούν με το συμβιβασμό και έτσι λοιπόν δεν μπορούν να τον υποστηρίξουν. Έχουμε την τεχνική που ακολουθούμε ως ήθιστε πάντα στην Επιτροπή μας. Τροπολογία 23 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτής. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 24. Συγγνώμη, μια στιγμή. Καταπίπτει αυτή. Η τροπολογία 25 τώρα. 25. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 26. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. ΔΕΒΕ 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. ΔΕΒΕ 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 28. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 29. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 30. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 1α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 32. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός 2. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 35. Άρχεται. Συγγνώμη, όχι. Εγκρίθηκε η προηγούμενη καταπίπτει αυτή. Τροπολογία ΔΕΒΕ 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 38. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε. Τροπολογία 37 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 39 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 3 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 4 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 42 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 43 πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα της ίδιας τροπολογίας 43. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε, τροπολογία 3 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε, τροπολογία 4 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε, τροπολογία 5 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε, τροπολογία 6 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 7 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 9 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 10 δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Ε, πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 11. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 13 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 4α. 4α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 15. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε. Τροπολογία 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18 πρώτο τμήμα άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 18 δεύτερο τμήμα άρχεται. Πέρας Εγκρίθηκε. Τροπολογία 19. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 19. 20 διορθώνει ο πρόεδρος. 20 φυσικά. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 22 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Θα ψηφίσουμε τώρα το σύνολο όπως τροποποιήθηκε της έκθεσης. Άρχεται. Πέρας. Με 21 ψήφους υπέρ και μία ψήφο εναντίον εγκρίθηκε. Καμία αποχή βέβαια. Συγχαρητήρια παρακαλώ στην κυρία Φράγκα. θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξή μας που είναι το σημείο 6. Ειδικοί όροι που αφορούν την από αποθεμάτων βαθαίων υδάτων στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό και διατάξεων που αφορούν την διεθνή αλληλεία στον Βορειοανατολικό Ατλαντικό καθώς και την κατάργηση του κανονισμού 2347 του 2002. Όπως γνωρίζετε είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων. Σχεδόν ε, για την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης που παρουσιάστηκε το Μάρτιο συνολικά καθορίστηκαν για τις 27 Μαρτίου οι ε, προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Θα έχουμε τώρα και μια ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες. Όπως πάντα πρώτα δίνω τον λόγο στον ίδιο τον εισηγητή, τον κύριο εισηγητή. Παρακαλώ. Gracias, Presidente. Thank you very much. Maybe we should... Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, ε, να τακτοποιηθούν λίγο οι συνάδελφοι μετά την ε, ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Έχουμε πάνω από 300 τροπολογίες, συγκεκριμένε 345 ε, τροπολογίες που αφορούν σε αυτήν την έκθεση. Εκφράστηκαν πολλές απόψεις για διάφορα θέματα και αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο περιθώριο για να επιτευχθεί συμβασμό σε αυτήν την Επιτροπή. Έχουμε εξετάσει όλες τις τροπολογίες ε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Χριστίνα και εγώ ε, συνεργαστήκαμε για να καταλήξουμε στο πακέτο του συμβιβασμού ε, αυτό. Το παρουσιάσουμε στην πρώτη συνάντηση με τους και ηγητές και έχουμε το δεύτερο πακέτο το οποίο περιλαμβάνει τα πιο περίπλοκα στοιχεία του άρθρου 9 αλλά και άλλα θέματα που αφορούν στην απαγόρευση. Και αυτά τα παρουσιάσαμε. Επίσης, η συνάντηση των ε, συντονιστών ε, έχει επιληφθεί του να αναζητήσει και αυτοί συμβιβασμούς. Όπως ξέρετε, είμαι ανοιχτός ε, για να υπάρξουν διαβουλεύσεις ε, με τη βιομηχανία αλλά και με πολλούς άλλους. Και οι περισσότεροι από εσά έχουν δει και την επιστολή ε, που έστειλε ο κλάδος και εκεί γίνονται σχόλια για διάφορες τροπολογίες. Μιλάμε λοιπόν με όλους και προσπαθούμε να βρούμε τις βέλτιστες δυνατές συμβαστικές λύσεις. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε από τις τροπολογίες των συναντέλφων αλλά και από τις συζητήσεις με τους σκιώδεις είναι ότι παρότι υπάρχει διάσταση απόψεων σε θέματα που αφορούν κυρίως στην απαγόρευση δηλαδή ε, στην απαγόρευση ε, στο ότι σιγά σιγά εκπνέει η απαγόρευση των τρατών ε, βαθέων υδάτων. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε λιγάκι τις ε, συζητήσεις. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι Είμαι αισιόδοξο. Μοιάζει ε, να πρόκειται να επιτεθεί ένα ευρύτερο πακέτο σε αυτήν την Επιτροπή. Είμαι αισιόδοξο, όπω είπα. Ε, τον Οκτώβρη νομίζω ε, θα καταλήξουμε τελικά σε μια ουσιαστική έκθεση. Και όπως πάντα και το γραφείο μου και εγώ είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις ή θέματα που θέλετε να συζητήσετε. Είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία αυτή που ε, προσπαθούμε να εγκαινιάσουμε. Δεν μιλάμε μόνο με ε, ε, τον αλληλευτικό κλάδο, αλλά ενδιαφερόμαστε για τα συμφέροντα όλων των κρατών που εκπροσωπούνται εδώ. Τους συναντήσαμε και προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε ε, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλήξουμε σε συμφωνία στην Επιτροπή. Και πρέπει να σας πω, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι πολύ σύντομα θα καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία. Σα ευχαριστούμε, κύριε Βαλένσα. Δεν ήξερα ότι θα πήγαινε τόσο γρήγορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτός ο νέος κανονισμός για τα αλλιεύματα βαθέων υδάτων. Έχει φυσικά και κάποιους νομικούς κινδύνους που συνεπάγονται για τα κράτη-μέλη σε σχέση με ποσοστώσεις που ανταλλάσσονται με άλλα κράτη-μέλη. Αυτό σε σχέση με τη διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 5 για τον κανονισμό που προτείνεται προβλέπει μόνο εκείνα τα αλλιεύματα θα μπορούν να αλλιεύονται που προηγούμενα αλλιευόντουσαν. Δηλαδή εκείνα τα κράτη που είχαν, μια, είχαν μικρότερες ποσοστώσεις, ας το πω έτσι, τώρα εξαναγκάζονται να μεταθέσουν το την αλλιευτική προσπάθεια σε άλλες ποσοστώσεις. Και αυτό θα σημαίνει στο μέλλον πιθανόν απώλειες για αυτά. Και αυτό είναι μια παραβίαση της αρχής της σταθερότητας Περί πρόκειται. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν εχέγγυα μια εγγύηση ότι δηλαδή θα μπορούν επ' αυτού να αλλιεύουν τα αλλιεύματα βαθαίων υδάτων. Γι' αυτό θα ήθελα από κοινού με άλλους την τροπολογία μας την 104 και την 203 να επιστήσω την προσοχή επί του θέματος. Μια τέτοια εγγύηση για την εκμετάλλευση θα προβλέπει την ελάχιστη εκμετάλλευση που θα διασφαλίζεται σε ποσόστοση από αυτά τα κράτη. Τώρα, για άλλα κράτη, άσχετα από το αν είχαν αντίστοιχη αλλιευτική προσπάθεια ή όχι, θα πρέπει να διασφαλίζεται σε αυτά τα κράτη ότι οπωσδήποτε θα μπορούν να αλλιεύουν αυτά τα αλλιεύματα αν οικονομικά και ε, τεχνικά είναι εφικτό. Ευελπιστώ ότι η τροπολογία μου θα μπορέσει να οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σα Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον κύριο Αρσένη για το ανοιχτό πνεύμα που επέδειξε ε, στις ε, εισαγωγικές του παρατηρήσεις. Αλλά ειλικρινά είναι πάρα πολύ ανοιχτός και ήταν ατέλειωτες αυτές οι συναντήσεις που είχαμε για διαβουλεύσεις. Ε, μέχρι τώρα είχαμε και πάρα πολλές ε, ακροα στην Επιτροπή και πολλές ε, συναντήσεις κατηδίαν. Η πιο πρόσφατη οργανώθηκε από τον συνάδελφό μας Τόμας, μια συνάντηση που ήταν πάρα πολύ χρήσιμη, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνάντηση γιατί είχαμε τον, τον Πλάσλεν από το ICEs ο οποίος μας είπε ότι γίνεται αλήψη περίπου 70.000 τόνων των βασικών ειδών βαθέων υδάτων από το 2000 και τώρα μειώθηκε, μειώθηκαν τα λιεύματα σε 35.000 τόνους, δηλαδή κατά το ίμιση της, ε, του αρχικού και σιγά σιγά λέω ότι επιτυγχάνουμε το MSY στα βασικά είδη, ότι βελτιώνεται η βιομάζα. Αυτά ελέγχθησαν πριν από δύο εβδομάδες και κατόπιν έχουμε, είχαμε και τον Λοράν ε, Πασκάλ, ο οποίος ε, αναφέρθηκε στην αλία βαθέων υδάτων και λέει μάλιστα πιο συγκεκριμένα αναφέρεται σε απαγόρευση ε, της βαθιά των κάτω από τα 200 μέτρα θα ήταν ε, ανόητο γιατί επισημαίνει πως οι καρχαρίες ε, και άλλα είδη θα ήταν βάλωτα σε παραγάδια και είχαμε και μια συζήτηση με τους ειδικού του κλάδου που εκπροσωπούσαν τη Σκοτία ε, κυρίως τα λευκά είδη και πήραν και ένα, μια συγκεκριμένη διάκριση, ένα βραβείο. Και είπαν λοιπόν ότι τελικά αν απαγορεύσετε κάθε είδος αλίας βαθέων υδάτων, τότε πώς θα μπορούμε κι εμείς να πουλάμε αυτά τα σκάφη, αυτές τις τράτες. Γιατί αν απαγορευτούν σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα μπορούμε να πουλάμε πουθενά αυτά τα αλλιευτικά σκάφη. Και αν αυτό συμβεί πώς θα μπορούμε να ε, μετατρέψουμε τα σκάφη αυτά, τα σκάφη αυτά σε ε, σε παραγάδια, σε σκάφη με παραγάδια. Εσείς λοιπόν λέτε ότι πρέπει να προτείνουμε σε, μια, σε ένα συγκεκριμένο είδος αλίας να λαμβάνει χώρα μόνο με σκάφη που αλλιεύουν παραγάδια σε παρα, με παραγαδιάρικα σκάφη. Το θέμα είναι ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε συμβαστική πρόταση, γιατί το άρθρο 9 λέει ότι ανεξάρτητα με το τι θα συμφωνήσουμε σε αυτή την Επιτροπή, μετά από δύο χρόνια όλες οι άδειες ε, ε, αλίας βαθέων υδάτων θα αποσυρθούν Γι' αυτό λοιπόν, ε, γιατί χάνουμε χρόνο να μιλάμε για συμβαστικές προτάσεις τη στιγμή που το άρθρο 9 περιλαμβάνει αυτή την έννοια της απαγόρευσης μετά από δύο χρόνια. Ε, δεν ξέρω πού ακριβώς κατευθυνόμαστε, αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ ε, υπάρχουν λανθασμένες απόψεις. Οι επιστήμονες και το ICE λέει λένε κάτι συγκεκριμένο. Από την άλλη έχουμε βέβαια τις ΜΚΟ που είναι πολύ πιο ισχυρές γιατί αυτές και έχουν τεράστια χρήματα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο και αυτές οι ΜΚΟ μοιάζει να λένε κάτι λίγο διαφορετικό. Γι' αυτό λοιπόν ας τα ξεκαθαρίσουμε λιγάκι τα πράγματα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας και πάλι στον κύριο Αρσένη ότι η δουλειά του ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Σας ευχαριστούμε κύριε Στίβενσον. Η κυρία Φράγκα. καθώς είμαι σκιώδης εισηγήτρια, εισηγήτρια και διαπραγματεύομαι και με τον κύριο Ασένη και τις σκιώδη εισηγητές, ε, εδώ πρέπει να διαρωτηθούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Όπως ξέρει ο κύριος Αρσένης και δημόσια αναφέρθηκε και αυτό το οποίο ε, ανέφερε ο κύριος Στίβενσον. Για μας υπάρχει ένα σημείο θεμελιώδου σημασίας που είναι το άρθρο 9 και είμαστε κατά κάθετα της πρόβλεψης οποιοδήποτε facing out σχετικά με αυτό. Είναι ένα άρθρο που δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε και συνδέεται με το άρθρο 9, το 4. Και γι' αυτό λοιπόν αυτή είναι η ουσία, ο πυρήνας της πρότασης. Τα υπόλοιπα όλα, τα υπόλοιπα Προφανώς υπάρχουν σαφείς τροπολογίες όπου γίνεται λόγος για ε, ζώνες αλλιές, νέες ζώνες, ε, διαφοροποιούμενες σημεία από την άλλη κτλ. κτλ. Και όπως έχουμε τις ε, τροπολογίες, εξοικονομώ το να σχολιάσω επ' αυτών. Αλλά φυσικά τα ουσιώδη σημεία είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν και να αποσαφηνίσουμε με τον κύριο Ασένη και από αυτό ως εκκίνηση τα υπόλοιπα είναι διαπραγματεύσιμα και μπορούμε να βρούμε τρόπους που θα ικανοποιούν αμφότερες τις πλευρές, λύσεις που θα ικανοποιούν αμφότερους. Για το άρθρο 9 Πρόκειται για μια πρόταση απόλυτα ριζοσπαστική αυτή που υποβάλλεται και δεν είναι ισορροπημένη και γι' αυτό εξακολουθώ να λέω ότι είναι ένα άρθρο το οποίο δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Μια και οι επιστήμονες, ε, οι περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας κτλ. ακολουθούν διαφορετικές οδούς για να μην αναφέρω τα Ηνωμένα Έθνη, τον ΦΑΟ λοιπά, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων. Μια πρόταση λοιπόν που θα έχει την ε, ίδια επικέντρωση, χωρίς να υπάρχουν ε, επιζήμιες επιπτώσεις ε, και αν έχουμε μια πιο σωστή επικέντρωση όσον αφορά τη διασφάλιση του ευάλωτου θαλάσσιου οικοσυστήματος, αυτό πιστεύουμε ότι είναι η σωστή πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Τώρα για τον κύριο Ασένη και πάλι υπέρ αυτού, διότι έχει μια διαφορετική πρόταση σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό είναι το σωστό. Διαπραγματευόμαστε με τον κύριο Αρσένη και φυσικά σε ένα πλαίσιο διαλόγου για το οποίο ευχαριστώ συνεργαζόμαστε με τον κύριο Αρσένη λέγοντας ποια είναι τα σημεία τα οποία αφορούν συμβιβασμούς και μπορούν να γίνουν ή όχι αποδεκτά και Και φυσικά τώρα Έχουμε και το, τη δέσμη προτάσεων, όπως είπα για το, άρθρο, για, το 4, για το άρθρο 4 και το 9, που είναι ουσιαστικά σημεία, πρέπει να δούμε ποια συμφωνία θα επιτευχθεί από αυτόν και πιστεύω ότι βρισκόμαστε όλοι απόλυτα πρόθυμοι στο να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο συμβιβασμό, ακολουθώντας μια γραμμή ευθυγραμμισμένη με ισορροπημένες προτάσεις και όχι με μια ε, πορεία που δεν θα οδηγεί σε μια ευσταθή και ισορροπημένη πρόταση. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό το οποίο επιθυμεί εξάλλου ο κύριο Ασέντη και το οποίο θέλουμε και εμείς. Πρέπει να συμβιβαστούμε και να καταλήξουμε σε ένα σημείο συνάντηση, σε ένα σημείο σύμπτωση απόψεων, ώστε να καταφέρουμε με τον κύριο Ασένη να επιτύχουμε αυτό το στόχο που έχουμε ενώπιόν μα και θέλουμε να διασφαλίσουμε. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιπε τροπολογίε μα είναι σε ένα σαφέ ε, πλαίσιο προτάσεων, ισορροπημένε και, και ε, ε, είναι θεμητό αυτό και έτσι λοιπόν ναι, για τα σημεία τα οποία θεώρησα σημαντικά σε αυτά αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς κυρία έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τις γνώσεις και την σοφία του εισηγητή που κατάλαβε τη σημασία και τις επιπτώσεις που θα έχει ο κανονισμός σε πολλές χώρες της Ένωσης και σε εκατοντάδες αλλιευτικά πλοιάρια. Και γι' αυτό θέλησε να κάνει πολλές συνεννοήσεις, όπως απαιτούνταν εξάλλου. Σήμερα δεν υπάρχει βέβαια συμβιβασμός, ιδιαίτερα ως προς τις απαγορεύσεις της στράτας, ούτε καν προοδευτική απαγόρευση. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοιο συμβιβασμό και ο μόνος πιθανός και δυνατός συμβιβασμό αφορά την μερική απαγόρευση, δηλαδή αναγεωγραφική ζώνη αλλά όχι στο σύνολο των βαθέων υδάτων που αλλιεύονται. Η ριζοσπαστική πρόταση θα ήταν η ολοκληρωτική απαγόρευση ακόμα και αν γίνει προοδευτικά. Το θέμα όμως είναι με τι όρους. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όχι για την πλήρη απαγόρευση αλλά για την απαγόρευση αναζώνες με βάση τις περιβαλλοντολογικές συνέπειες και μια συνεπή χαρτογράφηση. Γιατί υπάρχουν είδη βυθού που πρέπει να προστατευθούν, υπάρχουν οι ζηματικοί βυθοί που δεν έχουν πρόβλημα και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε να πούμε ότι δεν χρειάζεται και η απαγόρευση. Νομίζω λοιπόν ότι με βάση μια σοβαρή χαρτογράφηση και κατανομή αναζώνες θα μπορούσα να φανταστώ ως συμβιβασμό αυτή τη μερική επαναζώνες απαγόρευση. Φαντάζομαι ότι δεν θα επιτευχθεί εύκολα γιατί έχουν και οι μεν και οι δε πολύ επίμονες θέσεις, αλλά αν επιμείνουμε νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί ο συμβιβασμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Καντέκ. Oui, merci, monsieur le président. D'abord, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και τους σκιώδης και ευχαριστώ και την Κάρμεν που δέχτηκε να γίνει σκιώδης εδώ γιατί και εγώ έχω ασχοληθεί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλίας επί το οποίο θα χρειαστεί να ψηφίσουμε σε λίγες εβδομάδες και γι' αυτό ζήτησα από την Κάρμεν η οποία ευγενώς το δέχτηκε να γίνει σκιώδης. Ενδιαφέρομαι και εγώ βέβαια για το θέμα. Είναι εξάλλου σημαντικό να διαπιστώσουμε ότι έχουν κατατεθεί πολλές τροπολογίες, το είπε και ο Κρήτον. Και ότι υπάρχουν πολλοί στεναρές και διαφοροποιημένες απόψεις, το είπε και η Κάρμεν. Επομένως οι πιθανοί συμβιβασμοί που είναι απαραίτητοι θα είναι δύσκολοι. Ο συνάδελφός μας Κρήτον φαίνεται αισιόδοξο ως προς την επίτευξη των συμβιβασμών, εγώ είμαι λιγότερο αισιόδοξο. Α, θα δούμε, θα δούμε. Πάντως θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η θέση μου επί του θέματος αυτού. όπως είπε και η Σαβέλα Θωμά, η πλήρης απαγόρευση των σειρωμένων δικτύων μάλλον δεν θα επιτευχθεί. Οι αλληλείς θα μπορούν να ψαρεύουν σε ορισμένες ζώνες που έχουν γίνει αποδεκτές και έτσι θα δημιουργηθούν ζώνες αναδημιουργίας του αποθέματος. Όπως εξάλλου έλεγε και ο συνάδελφος Μιλάνα που δεν έχει απόλυτα άδικο. Οι ζώνες λοιπόν αυτές μερικής απαγόρευσης θα επιτρέψουν την αναδημιουργία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Έξω, πέρα από τις παγωμένες τελείως ζώνες. Λοιπόν, για τις σε εισαγωγικά δανεικές αυτές ζώνες έχω συζητήσει με επιχειρήσεις και μου είπαν ότι Όταν ψαρεύουν οι τράτες επί χιλιόμετρα στην ίδια γραμμή είναι σαν να πηγαίνουν βόλτα το σκύλο τους. Και συμφωνώ εδώ με την Κάρμεν Φράγα και την Σαμπέλ Τωμά ότι μία πλήρης απαγόρευση όπως προτείνει το σημείο 5 που είναι πολύ ριζοπαστική είναι απαράδεκτη και δεν θα οδηγήσει πουθενά. Και ε, ίσως να καταδικάσει πλήρως το είδος αυτό αλλιές που είναι το πιο διαδεδομένο κατά μήκο των ακτών μας. Εξάλλου δεν είναι στόχος της ε, Κομισιόν αυτή η πλήρης απαγόρευση. Εγώ βέβαια δεν έχω πιστεί για όλα αυτά και είτε το πιστεύει κανείς όμως είτε όχι θα δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για την αλληλεία με τα μέτρα αυτά. Αυτό να μην το ξεχνάμε μπορούμε να δεχτούμε το άρθρο 9 και το 4 και το 4 της Κομισιόν που το υποστηρίζει και ο Κρήτον Αρσένης γενικά. Επίσης εγώ θα ήθελα να μιλήσω για ορισμένες αρχές, δηλαδή πρέπει να υπάρξουν μέτρα διαχείρισης που πρότεινε η ΝΑΦΚ, το είπε και η Κάρμεν. Επίσης σημαντικό είναι να διαχωρίσουμε τα στοχευμένα ήδη από τα μη στοχευμένα, να υπάρξουν ανώτατα όρια για να υπάρξει και σωστότερη διαχείριση και δεν πρέπει να μείνουμε στα αυστηρά πολιτικά πλαίσια. Υπάρχουν και τεχνικά θέματα που πρέπει να λύσουμε. Άρχισε εξάλλου να το συζητάμε αυτό το θέμα η συνάντηση των σκιωδών. Να είναι μέτρα εφαρμόσιμα που να επιτρέπουν τη συνέχιση της αλλιευτικής δραστηριότητας. Επίσης Νομίζω ότι ο αυστηρός έλεγχος της αλληλείας αυτής είναι επίσης ουσιώδης για να διατηρηθούν τα ευαίσθητα είδη, όλοι συμφωνούμε γι' αυτό, να σεβαστούμε τα ανώτατα βιώσιμα επίπεδα αλίευσης και την αρχή της φρόνησης. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε και γι' αυτό το 9 και το 4 εντάξει υπάρχουν διαφωνίες, μπορεί να υπάρξουν και συμβιβασμοί αλλά δεν είναι σίγουρο. Ευχαριστώ κύριε Δρομέβα. Ευχαριστώ. Uh, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά που έκανε ο συγητής μας, διότι εδώ πρόκειται για κάτι που είναι και δύσκολο και δείχνει με απόλυτη σαφήνεια ότι υπάρχουν δύο ξεκάθαρες γραμμές. Αρκεί να διαβάσει κανείς τις ε, τροπολογίες για να δει ότι υπάρχουν δύο δυνατότητες για να προσεγγίσει κανείς τη συζήτηση. Τουλάχιστον κάτω έτσι από διεθνές ε, πρίσμα, κάπως γενικότερα δηλαδή. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να έχει κανείς ε, μια εικόνα της κατάστασης. Και θέλω να απαντήσω στον συνάδελφο Στίβενσον, ο οποίος αμφισβητεί το ρόλο των ΜΚΟ. Είναι σαφές ότι τα αποθέματα κινδυνεύουν. Και η αλία δεν γίνεται με βιώσιμο τρόπο. Αυτό το λέει η επιστήμη, δεν το λέει ναι, η ΜΚΟ. Η ΜΚΟ το εκμεταλλεύονται βέβαια. Αλλά το να τις κατηγορεί κανείς ότι αυτό λένε, αυτό είναι λάθος. Και πέρα από αυτό, θέλω να πω το εξής. Επιμένω σε τρία τουλάχιστον θέματα που η ομάδα μας επιθυμεί να υπάρχουν στο τελικό κείμενο. Θέλω να υπενθυμίσω... Μισό λεπτό κυρία Τόμας. Έχουμε λοιπόν τρία στοιχεία που θέλουμε να υπάρχουν στο τελικό κείμενο. Και υπάρχουν και τρία βήματα. Το ένα είναι η Επιτροπή, αλλά προβλέπεται και συγκεκριμένος ρόλος που διαδραματίζεται στην Ολομέλεια. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εδώ πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό και πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη θέση των συναδέλφων και εκτός αυτής της αίθουσας. Υπάρχουν λοιπόν τρία θέματα επί των οποίων έχουμε δεσμευτεί. Θα θέλαμε να υπάρχουν στο τέλος του κειμένου και ε, θέλουμε να υπάρξουν και ε, διαπραγματεύσεις για τις τροπολογίες. Ε, το ένα που είναι σημαντικό είναι το εξής. Ε, το ε, εξαφανιστούν οι μηχανότρατες κάτω από ένα συγκεκριμένο βάθος. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Είμαστε κατηγορηματικοί από αυτού. Βεβαίως μπορούμε λιγάκι να διαπραγματευτούμε το θέμα του ε, βάθους. Ίσως εκεί να βρούμε κάποια συμβαστική πρόταση. Αλλά είναι απόλυτα σαφές ότι θέλουμε να είμαστε σοβαροί στις προτάσεις μας. Άρα δηλαδή αυτό που σας λέω πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο τελικό κείμενο. Κατόπιν εδώ θέλω να προσθέσω κάτι και ίσως αυτό να ε, αφορά και αυτά που είπε η κυρία Φράγκα. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι να βασίζεται σε ε, τμηματικά μέτρα. Υπάρχουν τα ψηφίσματα ε, των Ηνωμένων Εθνών που πρέπει να είναι αυτά που μας καθοδηγούν. Γιατί λοιπόν να λάβουμε τμηματικά μέτρα τη στιγμή που μπορούμε να έχουμε μία παγκόσμια στάση με βάση τα ε, ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταστεί απόλυτα σαφές. Το ΝΙΕΦ ε, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι απαραίτητα ε, το βέλτιστο πλαίσιο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω οι του ευάλωτου δηλαδή θαλάσσιου περιβάλλοντος, του vulnerable marine environment. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν υπάρχουν ε, αρκετές ε, πληροφορίες, ε, χρειαζόμαστε καλύτερες αξιολογήσεις για τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε κάποιες περιοχές. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περιορίσουμε αυτές τις αξιολογήσεις μόνο στο αποτύπωμα. Δεν είναι σωστό αυτό. Ε, πρέπει να γίνονται αξιολογήσεις οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος και οπουδήποτε έχουμε ευάλωτο ε, θαλάσσιο ε, περιβάλλον. Και τέλος, κάτι άλλο, το οποίο είναι καθοριστική σημασία κατά την άποψή μας. Αν θέλετε, μπορούμε να διαπραγματευτούμε κάποιους όρους, αλλά όχι επί της αρχής δηλαδή τη μείωση αλληλευτικής ικανότητας ε, ε, στα είδη βαθέων υδάτων έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτά να αναπαραχθούν. Αν δεν συμφωνήσουμε επί της ουσίας της συζήτησης δεν νομίζω θα καταλήξουμε κάπου στο τέλος. Δηλαδή ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα αποθέματα να περιοριστούν ή να περιστεί η ελεκτική ικανότητα, αν δεν τα κατανοήσουμε όλα αυτά, τότε νομίζω ότι όλη η δουλειά θα είναι περιττή. Ο κύριος Στίβενσον μίλησε για το πόσο χρήσιμες είναι αυτές οι συζητήσεις και εγώ επίσης θέλω να πω ότι οι συζητήσεις θα είναι χρήσιμες ε, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θα προκύψει γιατί χρειαζόμαστε κάτι χρήσιμο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Επιστημονικά τουλάχιστον πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το πρόβλημα εφίσταται. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρωμέβα. Εσείς κύριε έχετε τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα είναι αυτονόητο και θέλω να ευχαριστήσω για την προσπάθεια που κατέβαλε ο εισηγητής κύριος Αρσένης. Διότι πιστεύω ότι πραγματικά από τις πρώτες συμβιβαστικές τροπολογίες που μας αποστάλησαν την Τετάρτη μέχρι το Σαββατοκύριακο υπάρχει πρόοδος στην πορεία και με τον απόλυτο σεβασμό για εκείνους που δεν τα γνωρίζουν όλα τέλεια και δεν τα έχουν αποσαφηνίσει όλα όπως σε τέτοια περίπλοκα θέματα όπως αυτά υπάρχουν τόσοι οικονομικοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, διαφορετικά συμφέροντα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ίδιας και άλλων πολλών ομάδων και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για τη μελέτη και την εξέτασή τους. Κυρίως επειδή υπάρχουν δύο δέσμες τροπολογιών. Υπάρχει μία δέσμη τροπολογιών που νόμιμα και με θεμητό τρόπο καταθέτουν κάποιοι ευρωβουλευτές. Εγώ δεν συμμετέχω επειδή ίσως ε, δεν με προσκάλεσαν σε αυτό αλλά είναι αυτονόητο και πρέπει να πω ότι παρότι δεν με προσκάλεσαν να συμμετάσχω σε αυτή την διαδικασία συμμετοχική και ευρύτερη όπου διάφοροι ευρωβουλευτές διαφορετικών πτερίγων του Κοινοβουλίου καταθέτουν τροπολογίες, τις ε, διαβάζω με προσοχή και βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες που συμπίπτουν επί της ουσίας με τις ίδιες τις τροπολογίες που εγώ ως ε, πλήρες μέλος ε, από την Ισπανική Αντιπροσωπεία για την Επιτροπή Αλλιέας συμφωνώ με αυτές, με άλλες δεν συμφωνώ. Υπάρχουν άλλες που είναι και αντιφατικές, αλλά έχουμε και το πακέτο συμβιβασμών, συμβαστικών τροπολογιών από την άλλη πλευρά, που αποκινούμε τις τροπολογίες πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια προσπάθεια για αυτές. Και προφανώς ε, αφουγκραζόμενοι και ακούγοντας ε, τις απόψεις των ε, διαφορετικών εμπλεκόμενων στον τομέα, στην Ισπανία για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προχωρήσει περισσότερο στη χαρτογραφία και στην μελέτη εξέταση αυτών των θεμάτων. Έχει γίνει μια δουλειά που έχει ξεκινήσει και που ουσιαστικά εδώ και ένα χρόνο καθορίζει με πολύ σε μεγάλη σαφήνεια τις ζώνες αυτές. Εδώ συζητώντας για τα είδη βαθαίων υδάτων ε, εδώ και γύρω από τις ε, παράκτιες περιοχές μας αυτό μας ε, αφορά άμεσα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε πολλά από τα, πολλές από τις στράτες που αλλιεύουν σε σχέση με, την... με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις υπό καμιά λοιπόν προϋπόθεση και μέχρι σήμερα τουλάχιστον θεωρώ ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό αν είμαι σωστά πληροφορημένη. Δεν υπάρχει ούτε ένα διεθνές φόρουμ ούτε στο ΟΗΕ, ούτε στην ΦΑΟ, ούτε αλλού που να έχει εξεταστεί η απαγόρευση αυτών των, τρατών. Άλλο θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε τώρα να βελτιώσουμε τους όρους προστασίας αυτών των ειδών σε σχέση με όλα τα μέσα τα επιστημονικά και τεχνολογικά και συμβουλές που μπορούν να μας διατεθούν από ε, τον επιστημονικό τομέα, από τους επιστήμονες για να αποφύγουμε την επιδίνωση του βιοτόπου, των βιοτόπων και να μην υπάρξει μια ας το πω έτσι, επιδείνωση των αλλιευμάτων που δεν θα μπορούν με να ανακάμψουν. Με αυτό το πνεύμα και αυτή τη φιλοσοφία που μας εμπνέει πρέπει να εργαστούμε. Εργαζόμενοι με αυστηρό και επιστημονικό τρόπο, χωρίς αυτό να, να μην αγνοήσουμε αυτό διότι δεν μπορεί να πολιτικοποιούνται τα θέματα και θα πρέπει κάποτε να ληφθούν αποφάσεις που πρέπει να είναι ισορροπημένες και κάθε ένας ε, έχει επιχειρήματα υπέρ χρησιμοποιώντας ε, τις απόψεις του που μπορεί να θεωρεί την οι πιο ορθολογικές. Ε, θα πρέπει να εισακουστούν όλες οι απόψεις βέβαια, αλλά πιστεύω ότι η βιασύνη σε, για αυτή την έκθεση δεν εξυπηρετεί κανέναν να εξευρεθεί, ας το πω έτσι, η γεφυροποίηση, η μέθοδος που θα δώσει δυνατότητα να συμβιβαστούμε και να βρούμε τον πιο ισορροπημένο τρόπο να πούμε ότι κάποια είδη πρέπει να απαγορεύονται απαγορευτούν οι διαλύες, πρέπει να καθοριστούν οι ζώνες, να δούμε ποιες ζώνες θα είναι αυτές όπου θα επιτρέπεται η αλία χωρίς να υπάρχει επιζήμια επίπτωση για ιδιαίτερα αλλιεύματα και μετά μια έκθεση πρέπει να έχει και κονδύλια τα οποία θα ε, ακολουθούν ε, τα συμπεράσματα και τις συστάσεις είχαμε σχεδόν την πλειοψηφία των μελών που είχαν ε, εγκρίνει τις προβλέψεις του, τις προοπτικές του Συμβουλίου, χωρίς να συγχέουμε λοιπόν τα θέματα, στο τέλος τέλος ε, θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε σε σχέση με διάφορες απόψεις το τι θέλουμε να κάνουμε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τις διαφορές που εξακολουθούν να είναι βαθιές ε, και παρεκκλίνουν η μία θέση από την άλλη. Να καταφέρουμε να βρούμε την δυνατότητα σύντομα να εγκρίνουμε συμβιβασμούς ε, και από πλευρά της ισπανικής αντιπροσωπείας και με την διακριτική ευχέρεια και ελευθερία που μου δίνει ας το πω έτσι ε, η, ίδια αυτή ενασχόλησή μου με αυτά τα θέματα, με τις τροπολογίες που καταθέτονται πρέπει να εξεταστούν τα θέματα τα οποία εξετάζουμε και να ληφθούν υπόψη από τους ε, μεν και τους δε. Να γνωρίζουμε γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη σε σχέση με την Ισπανική αντιπροσωπεία κάποια θέματα. Εξετάζουμε τα θέματα ώστε να υπάρξουν ισορροπημένες λύσεις, μέτρα ισορροπημένα. Οι μεταρρυθμίσεις να μην είναι μονόδρομος, να μην είναι μονής ε, ε, μονοβαρούς κατεύθυνσης. Να εξετάσουμε τα θέματα αυτά υπεύθυνα. Έχουμε την ευθύνη να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των οικονομιών μας και του αλλιευτικού τομέα για μας στην Ισπανία ο ελευτικός τομέας είναι πολύ σημαντικός. Έχουμε και το θεμητό, ε, την θεμητή μας θέση και το νόμιμο αίτημα είμαστε οι μεγαλύτεροι καταναλωτές και έχουμε το θεμητό και νόμιμο αίτημα να υπερασπιστούμε σε σχέση με την, ε, ε, τις, τις ΟΣΕΜ, κοινέ οργανώσεις αγοράς, τα θέματα των καταναλωτών. Να γνωρίζουμε γιατί και πώς μπορεί να αλλιεύεται ένα είδος δεν θέλουμε να ληφθούμε εμείς ξεχωριστά υπόψη. Όχι ότι επειδή εμεί λέμε ότι είμαστε πιο ευαίσθητοι από άλλους, εξαρτάται πού θέτει ο καθένας το επίκεντρο ως ε, ε, ε, εκπροσώπηση των συμφερόντων του. Πού τίθεται το επίκεντρο. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι και πάνω απ' όλα πρέπει να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία τέλεια. Ξεκινάμε από μια έκθεση που εκινεί με κάποιες κατευθύνσεις απαγορευτικές και σε σχέση με όλα αυτά θα πρέπει να δούμε ότι δυσχεραίνουν το πλαίσιο. Ο ίδιος ο εισηγητής θα πρέπει να είναι εκείνος που θα το κάνει θα έχει ευρύτερο φάσμα απόψεων, ένα ευρύτερο ορίζοντα για να εξετάσει και να δει αν μπορεί να δεχθεί άλλες απόψεις και να τις εντάξει στην πρότασή του για να μπορέσουμε προς όφελος όλων του συνόλου του αλλιευτικού τομέα και του περιβάλλοντος να δράσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Πατραονέβες παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένας μεγάλος αριθμός και γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομη για αυτά τα θέματα, διότι τα σημαντικότερα νομίζω αναφέρθηκαν. Θέλω να αναφέρω το γεγονός ότι πολλές από αυτές τις τροπολογίες αυτού του μεγάλου αριθμού που κατατέθηκαν έχουν, ας το πω έτσι, ε, οδηγήσει σε παρέκκληση και πιο οξύς θέσεις ε, πιο αυστηρές θέσεις και οι αποστάσεις που χωρίζουν τη μία άποψη από την άλλη έχουν αυξηθεί και σε σχέση με τις προηγούμενες ευκαιρίες που είχαμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα υπάρχει απόκληση απόψεων. Είναι αρνητική ας το πω έτσι η γραμμή εκκίνησης, ένα περίπλοκο και δύσκολο πλαίσιο αλλά πιστεύω ότι ο συγητής ο Κρήτον Ασένης υιοθέτησε ένα πνεύμα ευρύτερης συνεννόησης και διαλόγου που διευκόλυνσε αρκετά την αναζήτηση συμβιβαστικών λύσεων. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτό το θέμα είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο και σε σχέση με θέματα όπως αυτά πρέπει να τα εξετάζουμε και να τα προσεγγίζουμε από όλες τις πτυχές και τα πρίσματα ε, που εμπλέκονται στην αλληλεία. Κοινωνικό, ε, ε, άξονα περιβαλλοντικό, άξονα οικονομικό άξονα και την ανάγκη της προστασίας των οικοσυστημάτων θαλάσσιων, ε, ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Δεν θέλουμε να καταστρέψουμε με κανένα τρόπο εκείνο που στην, ε, επί της ουσίας είναι η μεγαλύτερη επένδυσή μας για το μέλλον μας. Και επίσης ε, και πρέπει να υπάρξει συνένεση επ' αυτού. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να υπάρξουν λύσεις που θα διευκολύνουν απλά κάποια πράγματα, θα είναι απλουστευτικές δεδομένων όλων των δυσκολιών και να μην είναι ισοπεδωτικές ε, οι προσεγγίσεις, να μην καταργούνται ή ακυρώνονται τα πάντα και ισοπεδώνουμε τα πράγματα με κάποιες ε, δράσεις μας. Και αυτή είναι μια πορεία που δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε λοιπόν. Αυτά που είδα σε σχέση με αυτήν την έκθεση είναι ότι ουσιαστικά πράγματι δημιουργήθηκε βήμα-βήμα σταδιακά ένα θετικό πνεύμα, ένα θετικός περίγυρος για να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας ημέν με τους δε. Και σε σχέση με συγκεκριμένα συμφέροντα των υπερπόντιων και υπερπεριφερειακών διαμερισμάτων και υπάρχει ευαισθησία σε σχέση με τον εισηγητή για αυτά τα θέματα και σε σχέση και με άλλα γενικότερα θέματα γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου που συμμερίζονται εξάλλου και ένα σημαντικό, συμμερίζεται ένα σημαντικό αριθμό ευρωβουλευτών αυτές τις, αυτά τα μελήματα τις ανησυχίες μου. Σε σχέση με όλα αυτά τα θέματα θα είναι πιστεύω εφικτό να βρούμε μια πορεία συνεννόησης, μια σωστή πορεία, ενδιάμεση, μέση, μέση οδό που θα διασφαλίζει, ας το πω έτσι, την υγεία για το παρόν και το μέλλον των ε, ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων και θα διασφαλίζουμε επίσης Εξίσου αυτά που είναι τα συμφέροντα από την άλλη πλευρά των αλλιέων μας, του αλλιευτικού μας ε, στόλου ή από, υπό το οικονομικό πρίσμα και το, τα συμφέροντα των ε, πληθυσμών μας που εμπλέκονται στις αλλιευτικές δραστηριότητες και κοινωνικά και οικονομικά. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση πραγματικά αποτελεσματική και βιώσιμη. Και γι' αυτό αυτό είναι το νόημα της παρέμβασής μου πέρα από ένα, μια ψήφο εμπιστοσύνης ε, για την πορεία που ακολουθούμε, διότι σε σχέση με αυτά τα θέματα είναι σαφής οι τοποθετήσεις μου και από προηγούμενες παρεμβάσεις και από τις τροπολογίες που κατέθεσα. Και πρέπει ίσως να υπενθυμίσουμε εδώ ότι πραγματικά μέσα σε αυτή την προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων θα πρέπει επίσης ε, να εκινήσουμε από ε, δράσεις και σε πολλές ε, ακροάσεις ε, είχαμε στοιχεία αξιόπιστα που μας παρουσιάστηκαν και έχουμε και αυτή την πορεία που προς το μέλλον πρέπει να διασφαλιστεί την ανάγκη να δημιουργήσουμε χώρους όπου σε αυτούς η αλλιευτική δραστηριότητα θα μπορεί να επιτρέπεται χωρίς να υπάρχει καταστροφή και επιδείνωση των ευάλωτων θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω ε, αυτής της ε, ας το πω έτσι δράσης ε, στην χαρτογράφηση και αποτύπωση ώστε να ξέρουμε επιστημονικά τι γίνεται, τι πρέπει να κάνουμε και μέχρι ποιου σημείου να δράσουμε. Αυτά ήταν ένα κοινό σημείο θα έλεγα στη θέση μας για την αλία. Βασιζόμαστε θεμελιών με τις ε, θέσεις μας, ε, πολιτικές θέσεις, σε επιστημονικά τεκμήρια και στοιχεία. Σε αυτά πρέπει να θεμελιωνόμαστε και να πορευόμαστε προς το μέλλον. Αυτή είναι η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θέλω να δώσω όμως ψήφο εμπιστοσύνης ε, προς τον εισηγητή μας και τους σκιώδους εισηγητές και σκιώδεις εισηγήτριες. Έτσι πρέπει να πορευτούμε μετά από την αρνητική κίνηση που ήταν μονοβαρής. Και μέσω συνένεσης να καταλήξουμε σε μια μέση οδό, ώστε αυτοί οι τρεις μεγάλοι πυλώνες, κυριότεροι πυλώνες ως άξονες, της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, να μπορέσουν να ε, ισορροπημένα να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Ρόντουστ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τον ε, Κρήτον Αρσένη διότι πιστεύω ότι η δουλειά του είναι πάρα πολύ δύσκολη, από τις πιο δύσκολες ε, που κλήθηκαμε να κάνουμε. Κλήθηκε να κάνει ακροβασίες, να περάσει από τη μία θέση στην άλλη. Ε, και μερικές φορές αποκόμισα και την εντύπωση ότι ε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ γιατί οι θέσει των ενδιαφερομένων ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε διάφορες απόψεις, η συζήτηση έγινε και πολιτική, πολλοί μίλησαν και για το ότι είναι θέμα στάση ζωής. Για μένα είναι θέμα αξιολόγησης ε, των στοιχείων. Έχουμε, λοιπόν, είχαμε κατά το παρελθόν δύο μεγάλες ακροάσεις και ακούσαμε ότι πάρα πολλοί επιστήμονες λένε ότι πρέπει να ταχθούμε με την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να επιδιώξουμε μακροπρόθεσμα την απόλυτη απαγόρευση. Επίσης, στο πλαίσιο των ακροάσεων ακούσαμε ότι όσον αφορά τα παρεπίμπτοντα αλλιεύματα, εκεί περιλαμβάνονται και ψάρια ηλικία 150 ετών και ακόμα μεγαλύτερη. Και αυτά θα καταστραφούν. Ακόμα και αν ε, δεν ε, επιτρέψουμε κάτι τέτοιο στο μέλλον με τους ε, κανόνες της κοινή ελληνικής πολιτικής, παρόλα αυτά φαίνεται θα αλλιεύονται και ψάρια που έχουν τεράστιο κύκλο ζωής. Επίσης ακούσαμε ότι ο βυθός χρειάζεται από 3.000 μέχρι 5.000 χρόνια έτσι ώστε να αποκαταστήσει ας πούμε τα κοραλιοφόρα πεδία γιατί ακούσαμε ότι υπάρχουν και βυθοί που δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Και εδώ θα είμαι πολύ επιθετική. Ίσως εμείς να φταίμε γι' αυτό. Γιατί κατά τα προηγούμενα ετή αναπτύξαμε δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν σε αυτούς τους βυθούς να αποκατασταθούν. Βέβαια δεν μου το είπε κανείς αυτό, εγώ ήθελα να είμαι επιθετική. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας γνωρίζουμε από την επιστήμη ότι και η επιστήμη σε πολλές περιπτώσεις σηκώνει ψηλά τα χέρια. Τα βαθαία ύδατα δεν έχουν τύχει τέτοιας μελέτης έτσι ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε αδιαμφισβήτητες απόψεις. Και λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι να πω δεν μπορώ να εκτιμήσω τις συνέπειες. Κατόπιν τούτου, όταν κληθώ να αποφασίσω ε, δεν μπορώ να αποφασίσω με βάση αυτό που είπε ο προηγούμενος συνάρφος ότι θα πρέπει και αυτοί που κατασκευάζουν τα παραγαδιάρικα να μπορούν να τα πουλήσουν. Ε, τι να πω κι εγώ, λυπάμαι πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, όταν καταστρέφεται ο βυθός ε, και η ελία βαθέων υδάτων, έτσι κι αλλιώς περιτά είναι τα παραγαδιάρικα. Τι να κάνουμε, λυπάμαι, αλλά πρέπει να το πω ξεκάθαρα και αυτό εμένα δεν θα με εμποδίσει να αποφασίσω αυτό που νομίζω. Όμως ε, την απόφασή μου θα την εξαρτήσω από αυτό που είπαν οι επιστήμονες με απόλυτη σαφήνεια εδώ στην αίθουσα και δεν άκουσα κανένα επιστήμονα που να μας είπε, ξέρετε, ε, αποφασίστε αυτό που θέλετε, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο τραγικά. Η δική μου η άποψη είναι αυτή που σας είπα, στην ομάδα εργασίας ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, αλλά σας λέω ήδη τώρα ότι επειδή υπάρχουν τόσες πολλές ασάφειες, εγώ δεν μπορώ να αποφασίσω ότι τα πράγματα θα συνεχιστούν ως έχουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή Κρήτονα Αρσένη για την εξαιρετική του εργασία. Και της Κομισιόν η δουλειά ήταν εξαιρετική και υποστηρίζω πλήρως αυτά που της υπόλοιπης επιτροπής μάλλον. Και υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπε και ο κύριος Ρωμέβα ένας από τους κοιόδης. Έχω προσέξει το θέμα αυτό αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι εκείνοι που θεωρούν ότι η επιστήμη θεωρεί ότι αυτού του είδους η αλληλεία είναι βιώσιμη, δεν ξέρω πού το βασίζουν. Γιατί εγώ καθ' όλες τις συζητήσεις πήγα στις ιστοσελίδες του ΆΙΣ και είδα ότι πολλά είδη ηχθείων είναι τελείως άγνωστοι οι τύχη τους και επομένως το μόνο που μπορούν να πούν οι επιστήμονες μέχρι τώρα είναι παρακαλώ αλλιεύετε τα λίγο λιγότερο. Και είπε και η κυρία Ρόντουστ ότι μερικά από αυτά τα είδη ε, είναι πολύ μακρόβια. Μερικά φτάνουν την ηλικία των 70 ετών και οριμάζουν σεξουαλικά στα 18 ή 18 τους χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για είδη που είναι πολύ ευπαθή. Αυτό είναι σαφές. Επίσης, για τι αλλιεύματα μιλάμε. 3.000-6.000 τόνοι. Συνάδελφοι, θυμηθείτε. Εδώ μιλάμε για 10.000 τόνους τι πράγματος ζωικής πρωτεΐνης για τροφή. Θέλουμε λοιπόν να καταστρέψουμε τελείως ορισμένα είδη για να τα φάμε. Σας υπενθυμίζω ότι του χρόνου στη θάλασσα του Μπάρεντς προβλέπεται η αλίευση ενός εκατομμυρίου τόνων βακαλάου. Γιατί θέλουμε λοιπόν συν 10.000 τόνους αγνώστων ειδών ηλικία της γιαγιάς σας. Δεν ξέρω αν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πετύχει πριν από μισό χρόνο να διαπραγματευτεί και να εγκρίνει μία βιώσιμη καινούργια κοινή αλλιευτική πολιτική και μας χειροκρότησαν οι ψηφοφόροι μας γιατί ο καθένας γνωρίζει ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής αλληλείας έχει καταλήξει σε καταστροφή των αποθεμάτων και αυτό αφορά όχι μόνο τη δική μας γενιά και τους τωρινούς αλληλείς αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Μας χειροκρότησαν λοιπόν γιατί λάβαμε υπεύθυνες αποφάσεις και αναρωτιέμαι τι μήνυμα στέλνουμε στους ψηφοφόρους μας εάν έξι μήνες αργότερα υπαναχωρήσουμε για να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα ενός πολύ μικρού τμήματος της αλληλευτικής δραστηριότητας ενώ όλοι συμφωνούν ότι είναι καταστροφική η δραστηριότητα η αλλίευση αυτών των ειδών. Νομίζω ότι θα δώσουμε μια εικόνα σχιζοφρένειας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανευθυνότητας και δεν νομίζω ότι αυτό θέλουμε να δείξουμε εν ώψη των ευρωεκλογών. Παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, η πρόταση της Κομισιόν είναι λογική νομίζω και όλες οι αξιολογήσεις που μας παρουσίασε ήταν πολύ προσεκτικές και ο αλληλευτικό τομέας δεν έχει καν αποφε... καταλήξει σε περισσότερα κέρδη από αυτού του είδους στην αλία. Παρακαλώ λοιπόν να συντομεύουμε τη διαδικασία, το έχουμε συζητήσει πολύ και ελπίζω να πάρουμε υπεύθυνες αποφάσεις. Σε ευχαριστώ κύριος Μιλάνα. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομα γιατί Πορά έχουν ήδη λεχθεί. Κοιτάξτε, και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια του κ. Σένη και τον ε, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά κάνει ε, ένα, μια εράκλεια προσπάθεια. Έχουν υποβληθεί τόσες ε, πολλές τροπολογίες και είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει κανείς και τους συσχετισμούς που αναπτύχθηκαν. Ευχαριστώ και τον κύριο Καντέκ, ο οποίος αισθάνεται, είναι, μοιάζει με τον Άγιο Παύλο όπως ε, λιθοβολήθηκε πηγαίνοντας στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Είναι λοιπόν ε, ίδια περίπου η κατάσταση. Εγώ πολύ ευχαρίστως ε, να μεσολαβήσω για να καταλήξουμε σε ένα συμβασμό και ίσως ε, τελικά να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ορισμένα σημεία. Θέλω επίσης ε, να πω ότι δεν ανησυχώ ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Και εκείνο που με απασχολεί είναι η σημασία που αποδίδεται στο ότι ξαφνικά πρέπει να πούμε σε κάποιον ότι δεν μπορεί πια να ψαρεύει. Και θέλω να επενθυμίσω σε όλους σας ότι όταν επρόκειτο για την κατάργηση της ε, άδειας ε, στα 3.000 μέτρα στη Μεσόγειο, τότε η Κομισιόν ήταν εκείνη που αποφάσισε και δεν ελήφθη κανένα μέτρο, κανένα αντίμετρο για αποζημίωση, για αποκατάσταση ή εν πάση περιπτώσει κάποια διαδικασία έτσι ώστε να υπάρξει κάποια ταύτιση ή κάποια κάλυψη των αναγκών του τομέα. Νομίζω λοιπόν πράγματι ότι μπορούμε, εγώ τουλάχιστον μπορώ να ε, διαμεσολαβήσω και προτείνω στον κύριο, Αρσένη, οποιαδήποτε μορφή διαμεσολάβηση. Αλλά τον παρακαλώ να μην καταπνίξει οτιδήποτε υπάρχει. Ναι, εντάξει, να ε, διαμεσολαβήσουμε, αλλά να μην μπούμε στην επιστημονική κοινότητα ότι είναι ομόφωνη η απόφαση. Κοιτάξτε, εδώ είμαστε ένα σημαντικό φορέας. Είμαστε η Επιτροπή Αλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά δεν είμαστε ομφαλός του κόσμου και, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε και ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Άρα, δηλαδή, καλό είναι να αναζητήσουμε κάποιες συμβαστικέ ε, προτάσεις, γιατί αν δεν υπάρξει πρόταση, τελικά αυτό θα ήταν πολύ κακό για όλου μα. Κακό για το δικό μας το ρόλο και κυρίως ε, αν δεν υπάρξει απόφαση τελικά δεν θα υπάρξει και διαμεσολάβηση. Θεωρώ λοιπόν ότι μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός και να το κάνουμε όλοι μας. Αν δεν υπάρξει διαμεσολάβηση όπως ε, σας είπα, αυτό κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά διότι ενδεχομένως να ακυρωθεί ο ρόλος μας. Και κλείνοντας, θέλω να κάνω μία πολύ απλή παρατήρηση. Να πω κάτι που έχει σχέση και με τα οικονομικής φύσεως θέματα. Να αναφερθώ λιγάκι στην αποδοτικότητα αυτού του τομέα. Κοιτάξτε, από την έκθεση ε, του ε, ελεγκτικού συνεδρίου της Γαλλίας του 2008 θυμάμαι ότι τα νέα αλλιευτικά σκάφη ε, στη Γαλλία επιδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το κράτος. Άρα δηλαδή η δραστηριότητα αυτών των σκαφών δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Και κλείνω λέγοντας το εξής. Δεν ξέρω κατά πόσον μία τράτα δεν μπορεί να ψαρέψει ίσως σε άλλα ύδατα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί και μάλιστα μπορεί να αναπροσαρμοστεί, να ανακατασκευαστεί. Αυτό που κάναμε και εμείς ε, σε άλλες περιπτώσεις. Και εν πάση περιπτώσει εγώ με πολύ μεγάλη χαρά να πω στον Κρήτονα να καταθέσει μια σύσταση στην Επιτροπή έτσι ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό τον κλάδο να συνοδεύεται και με άλλες ε, διατάξεις που θα την ενισχύουν. Δηλαδή τα σκάφη αυτά να μπορούν να ε, ανακατασκευάζονται και να χρησιμοποιούνται όχι σε βαθιά ύδατα αλλά σε άλλου είδους ύδατα. Yeah, thanks, uh, President. I... Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια, ένα σύντομο σχόλιο με βάση αυτά που είπε η κυρία Λίβινς. για τα ε, είδη που υποτίθεται ότι αφορά ο κανονισμός αυτός. Και σε ακροάσεις μάθαμε από εκπροσώπους των αλλιέων ότι μερικές φορές είχαν αντιμετωπίσει απρόβλεπτα αποτελέσματα προσπαθώντας να αλλιεύσουν ήδη βαθέων υδάτων. Και διαπιστώσαμε ότι οι επιχειρηματίες κυρίως ενδιαφέρονται για την αλίευση των ειδών αυτών και γι' αυτό θα έπρεπε ίσως να μετριάσουμε τις προτάσεις για να αποφευχθούν τέτοιου είδους απρόβλεπτες συνέπειες. Νομίζω ότι κατά την αναθεώρηση της ΚΑΛΠ ε, είχαμε εργαστεί πολύ λογικά και από ό,τι είχα καταλάβει εγώ είχαμε ζητήσει πιο αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων για να αντικατοπτρίζει περισσότερο την πραγματικότητα και δεν μιλούσαμε για πανευρωπαϊκές ε, ομοιόμορφες προτάσεις και γι' αυτό έχουν κατατεθεί ορισμένες τροπολογίες που επανέρχονται σε αυτά που είχαμε εγκρίνει για την αναθεώρηση της ΚΑΛΠ. για να μην καταργήσουμε έτσι μεγάλο τμήμα της κανονικής καθημερινής δραστηριότητας των ελιευτικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Έχω ζητήσει τον λόγο σε ένα δεύτερο γύρο κάποιοι ευρωβουλευτές που παρενέβησαν ήδη, καθώς ε, δεν πιέζει ιδιαίτερα ο χρόνος, θα το κάνουμε, αλλά πρώτα θα δώσουμε τον λόγο στην Επιτροπή, να τοποθετηθεί η Επιτροπή και μετά θα έχουμε ένα σύντομο δεύτερο γύρο. Και στο τέλος θα λέει τον λόγο ο εισηγητής κ. Αρσένης για να μας πει αυτά τα οποία θεωρεί ότι είναι αναγκαία να αναφέρει. Από την Επιτροπή εσείς παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει την Επιτροπή Ελίας μέχρι τώρα ε, με την έννοια ότι έχει προσφέρει διευκρινήσεις οπουδήποτε κρίθηκε αυτό απαραίτητο. Και ελπίζω να τα καταφέραμε. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την πρόοδο των διαβουλεύσεων και με μεγάλη μας χαρά να συνεχίσουμε να σας βοηθάμε αν αυτό ε, κριθεί απαραίτητο ε, για να επιτύχουμε το βασικό μας στόχο που είναι με στοχευμένο τρόπο να ε, επηρεάσουμε εκείνα τα ε, κυρίως που έχουν άμεση σχέση με τα βαθέα ύδατα. Η πρόταση της Επιτροπής ε, του να εξαλειφθούν ε, κάποια εργαλεία είναι μια στοχευμένη πρόταση. Να εξαλειφθούν κυρίως εκείνα τα οποία επηρεάζουν το περιβάλλον, όχι έτσι γενικά και όριστα. Ε, κατόπιν τούτου, με αυτή την έννοια της ε, στόχευσης, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες εκείνων που αναφέρονται στο να υπάρχει ένα όριο των 600 μέτρων διότι αν δει κανεί ε, τα βάθη ε, στα οποία γίνεται η αλεία μπορεί ε, να γίνεται αλεία αρκετών εμπορικών ειδών, τα οποία αναμφίβολα είναι εκτός του περιβάλλοντος βαθιών υδάτων, το οποίο ψάχνουμε. Πολλά είδη ψαριών μπορούν να τύχουν αλίες σε αυτό το βάθος, ε, άρα δηλαδή η γενίκευση ε, δεν είναι κάτι που επιθυμούμε. Θέλουμε όμως να πούμε ότι κάποια εργαλεία μπορούν να είναι επικίνδυνα, γι' αυτό θα πρέπει να ε, χρησιμοποιούνται με προσεκτικό τρόπο. Άρθρο 9 παραδείγματος χάρη. Αυτό αξίζει τον κόπο να το σκεφτούμε. Όπως σας είπα και στην αρχή, με μεγάλη μας χαρά ε, να βοηθήσουμε αν αυτό βοηθήσει την Επιτροπή. Και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα τα οποία συζητούνται και δεν θέλω να δαπανίσω το χρόνο σας για να μπω σε λεπτομέρειες. Αλλά ίσως μπορείτε να μου επιτρέψετε να τίξω ένα συγκεκριμένο θέμα, διότι ε, μπορούμε να υποφεληθούμε σε αυτό και από πράγματα που έχουμε μάθει σε άλλες μορφές αλίας. Υπάρχει μία πρόταση που λέει ότι παράλληλα με την, ε, όσον αφορά τη διαχείριση της αλίας βαθαίων θα πρέπει παράλληλα με τα μέγιστα αλευτικά θέματα, τα ΤΑΚ, να έχουμε και την αλευτική προσπάθεια. Ας πούμε, ξέρουμε όσον αφορά τον μπακαλιάρο στη Βόρεια Θάλασσα, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρχουν και τα δύο παράλληλα. Είναι πολύ χρήσιμα τα εργαλεία αυτά, αλλά ε, νομίζω ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να επιλέξει κανείς ε, μία από αυτές τις δραστηριότητες, αντί να τις αφήσει να συνεπάρχουν παράλληλα. Αυτά είχα να σας πω. Ε, να υπάρχει λοιπόν στοχευμένη συζήτηση και αν εμεί μπορούμε να βοηθήσουμε, παρακαλώ με μεγάλη μα χαρά θα το κάνουμε. Πολύ καλά, σα ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο γύρο. Παρακαλώ να είστε πιο σύντομοι. Η κυρία Φράγκα πρώτη, παρακαλώ. Ναι. Άκουσα τόσα πράγματα και εν πάση περιπτώσει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε σύντομοι. Να απαντήσω στον κύριο Ρουέβα σε αυτά που είπε για τα θέματα της βαθυμετρίας. Πρέπει επίσης να πω ότι σε σχέση με τον συγητή σε μια συμβιβαστική τροπολογία στο άρθρο 4 που συνδέεται με το άρθρο 9 συμπεριλαμβάνονται τα σκάφη που αλλιεύουν κάτω από βάθος 600 μέτρων. Το θέμα της βαθυμετρίας λοιπόν δεν είναι ένας ε, ε, συντελεστή που μπορεί να λαμβάνεται υπόψη με το σωστότερο τρόπο. Αν πούμε ότι σε χ ε, βάθος, ε, παράδειγμα 600 μέτρα, ε, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν άλλα είδη τα οποία βρίσκονται στα 400 μέτρα, τα οποία δεν θα προστατεύαμε. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αμμώδει βυθοί πυθμένε κάτω από 600, τα 600 μέτρα. Και τώρα να δούμε τι θα γίνεται σε σχέση με τις τράτες ε, ε, βαθέων υδάτων. Το θέμα της βαθυμετρίας δεν είναι το πιο σκόπιμο. Οι Νορβηγοί έχουν απαγορεύσει κάτω από 1500 μέτρα αυτή τη χρήση. Βλέπουμε εδώ τη διαφορά για τα 600 μέτρα που είναι μια πρόταση για παράδειγμα που δεν έχει κανένα νόημα σε σχέση με αυτό το βάθος. Αυτά που ανέφερε η κυρία Λεβίν για τα είδη, τα λιεύματα των βαθέων υδάτων για τις ε, μοιραίες επιπτώσεις ε, και ότι υπάρχει ε, η μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής και για το χρόνο που πρέπει να λάβουμε το μεγαλύτερο μέρος των ειδών για την ανάκαμψή τους όπως είναι διάφορα είδη πρέπει να υπάρξει, αν υπάρξει μείωση αλλιευτικής προσπάθειας στα 30% για τον κοινοτικό στόλο να μην μας λένε ότι όλα τα είδη των βαθέων υδάτων βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όλα και ε, ε, επιμένω επ' αυτού για το ε, μηδενικό επίπεδο. Είναι ένα είδος απαγόρευσης αυτό και πιστεύω ότι εδώ οι επιστήμονες έχουν διαφορετικές απόψεις από τα όσα λέγονται εδώ. Τα είδη βαθέων υδατών γενικά ανακάμπτουν, σημειώνουν ανάκαμψη και υπάρχουν μόνο κάποια είδη τα οποία βρίσκονται σε μια κατάσταση που έχει επιδεινωθεί και η πλειοψηφία τους δεν έχει αυτό το προσδόκιμο ζωής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας αναφέρετε. Εδώ και τις παρεμβάσεις που ακούω και μάλιστα από την αρχή αυτής της συζήτησης ακούω παρεμβάσεις ε, και τοποθετήσεις στις οποίες ουσιαστικά κατανοεί κανείς ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε και αναφερόμαστε σε επιστημονικά συμβούλια, επιστημονικές συμβουλές, παρότι το επιστημονικό συμβούλιο, και έχω εδώ για παράδειγμα τα στοιχεία, πρόκειται για τη σύνοψη της αντίστοιχης έκθεσης ε, του Γαλλικού Ιδρολογικού ε, Ιδρύματος, Ινστιτούτου. Έχει δημοσιευθεί και μόνο στα γαλλικά έχω αυτά τα στοιχεία. Σας συνιστώ θερμά να διαβάσετε αυτά τα συμπεράσματα και συστάσεις, διότι εξοργίζομαι όταν γίνεται λόγο εδώ για επιστημονικές απόψεις, επιστημονικά τεκμήρια, τα οποία είναι ανύπαρκτα. Δεν είναι δεδομένα όλα αυτά. Έχουμε ακροάσεις ε, με επιστήμονες που έγιναν εδώ και προσήλθαν οι επιστήμονες εδώ για να μας δώσουν αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να πω αυτό το άρθρο. Όλο το επιστημονικό ίδρυμα το υποστηρίζει, όλοι οι επιστήμονες που εργάζονται εκεί έχουν συμμετάσχει και λένε πρώτον για το βάθος για τα βαθαία ύδατα. Είναι ένας ορισμός, λέγεται, που καθορίζει αποκλειστικά μόνο το βάθος. Αν ένας τέτοιος ορισμός βασιζόταν μόνο σε συγκεκριμένο βάθος, τότε θα έπρεπε να αναφέρεται και στην ε, ε, υφαλοκρηπίδα και να αναφερόμαστε ε, σε σχέση με τα όρια υφαλοκρηπίδας μέχρι συγκεκριμένου βάθους και σε σχέση και με την φύση των παράπλευρων αλλιευμάτων. Τι γίνεται εδώ. Δεν σας τα διαβάζω όλα αυτού του άρθρου. Λέει όμως υπάρχουν παράπλευρα αλλιεύματα. Οι απορρίψεις παράπλευρων αλλιευμάτων έχουμε ε, δύο είδη που αφορώνται άμεσα, ε, καμιά φορά και ένα τρίτο είδος, για τα οποία όμως ε, δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση για την διασφάλιση της ανάκαμψης των αλλιευμάτων του και για τον έλεγχο της αλίας. Είναι ο πιο αυστηρά ελεγχόμενος τομέας αλίας. Υπάρχουν και επόπτες οι οποίοι βρίσκονται πολλές φορές στα ίδια τα σκάφη. Άλλες φορές δορυφορικά διασφαλίζεται η εποπτεία, η επιτήρηση. Για να γνωρίζουμε ακριβώς και να μπορούμε να γνωρίζουμε ποιο σκάφος που αλίευει και ποιου είδους αλιεύματα είναι αυτά που συλλαμβάνει. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να πούμε και αυτή η πτυχή εξίσου διασφαλίζεται. Τώρα για το RMD για τη διάγνωση και τις ε, γνωμοδοτήσεις από πλευράς 2012 όσον αφορά το πλαίσιο της επιστήμης. Οι επιστήμονες αναγνωρίζουν ότι η εκμετάλλευση των ειδών βαθέων υδάτων έχει επιτύχει ένα επίπεδο ανάκαμψης μετά την υπεραλίευση κατά την αρχή του 21ου αιώνα. Τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν ήταν θετικά και οδήγησαν σε μία ανάκαμψη των αλλιευμάτων. Ε, γοργά έγινε αυτό αισθητό από πλευράς ανάκαμψης που σημειώθηκε και για τα είδη βαθαίων υδάτων. Ε, αναφέρατε μας εσείς τώρα ποια είναι τα επιστημονικά συμπεράσματα στα οποία εσείς βασίζεστε. Έχω εδώ αυτά τα στοιχεία, τα έφερα εδώ, τα βλέπετε, να τα, πάρτε τα κι εσείς ε, να τα συμβουλευτείτε. Τα έχω μόνο στα γαλλικά βέβαια. Αν θέλετε στα αγγλικά να μεταφραστούν, ευχαρίστω να το κάνω προσωπικά, εγώ να σα τα μεταφράσω, παρότι δεν είναι τα πιο τέλεια τα αγγλικά μου. Δεν υπάρχει υπάρχει άλλη παρέμβαση. Ο κύριος Αρσένης είναι νυφάλιος. Έχετε τον λόγο κύριε Αρσένη. Uh, Κοιτάξτε, γνωρίζω το περιεχόμενο αυτού του κειμένου. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις ε, επιστημονικές απόψεις και είμαι εδώ για να καταλήξουμε σε κοινό παρονομαστή. Βεβαίω κοινό παρανομαστή σημαίνει ότι καταλήγουμε σε κάτι το οποίο έχει νόημα και ελπίζω να το πετύχουμε αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Έχουμε και είχαμε πολύ καλή δουλειά. Κάποια στιγμή θα την ολοκληρώσουμε. Ελπίζω να υπάρξει σύγκληση απόψεων στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι, ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Περνάμε στο επόμενο σημείο που είναι το 7. Πολιετέ ε, πρόγραμμα ανάκαμψη για τον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο για τον Ερυθρόπτερο Τόνο. Έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την παρουσίαση της πρότασής της ε, και στη συνέχεια φυσικά θα έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων. Από πλευρά τη Επιτροπής έχετε το λόγο εσείς κύριε Ντοματέλα παρακαλώ. Thank you, Chair. Sorry for this delay. Trying to find a place. Um, this proposal uh, reflects the decision. Εδώ αντικατοπτρίζεται η άποψη του ΣΚΙ σχετικά με την αποκατάσταση του ερυθρού τόνου. Μία από τις δυνατότητες που συζητήθηκε ήταν να προσαρμοστεί η αλευτική περίοδος για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές που υπάρχουν στα αλευτικά σκάφη αλλά και για να ληφθεί υπόψη ένα βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει ο τομέας ε, και δεν μιλάω για τον ευρωπαϊκό αλληλεκτικό τομέα, αλλά μιλάω και για άλλους τομείς έτσι ώστε να ληφθεί απολύτως υπόψη, να ληφθεί μία απόφαση έτσι ώστε να περιοριστεί η συγκεκριμένη αλληλευτική περίοδος έτσι ώστε να υπάρχει και αποκατάσταση του ερυθρού Αυτή λοιπόν η συζήτηση γίνεται με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους του κλάδου έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσον οι αλλαγές θα λαμβάνονται υπόψη ως μια επιπρόσθετη προσπάθεια ή να διαπιστωθεί κατά πόσο εκείνο που ενδιέφερε ήταν να δοθούν στον κλάδο τα εργαλεία έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητες που υπάρχουν στο πλαίσιο του σχεδίου ICAT και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών. Η πρόταση αυτή έχει σχέση με την τροποποίηση των σημαντικών διατάξεων που συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό 302 και ε, προ, περιλήφθηκαν αργότερα σε ένα μεταγενέστερο καορισμό. Έτσι λοιπόν ορίστηκε η αλληλευτική περίοδος ε, για πολλά σκάφη όπως ε, για τα παρακαδιάρικα αλλά και για τα ε, θυναλιευτικά και τα σκάφη ή τα γρηγρή. Πράγματι λοιπόν αυτή η συζήτηση που επικράτησε ήταν σχετικά με την αλληλευτική περίοδο. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι ότι αντί να υπάρχει μια κλειστή περίοδος, κάτι που δεν είναι απόλυτα σαφές για ορισμένα από τα συμβαλόμενα μέρη, συμφωνήσαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να υπάρχει σαφής ε, άποψη για το πότε μπορεί να ισχύει η αλληλευτική περίοδος, να διευκρινιστεί ε, για όλα τα λιευτικά σκάφη που αλλιεύουν τον ε, ερυθρό τόνο να ε, ισχύει περίοδος χωρίς περιορισμούς. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα λιευτικά σκάφη για να μπορούν να πτύξουν δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ βέβαια εκκρεμεί η εφαρμογή της νέα σύστασης που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2012 και θεωρούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τα πιο αυστηρά μέτρα. Και γι' αυτό τον λόγο σήμερα έχετε μπροστά σας αυτό το συγκεκριμένο θέμα που αφορά στο πρόγραμμα αποκατάστασης ε, του ερυθρού τόνου του Ατλαντικού. Βεβαίως, ε, σύντομα θα καταθέσουμε και άλλη μια πρόταση, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη και όλες οι άλλες ε, τροποποιήσεις που έχουν σχέση με τον έλεγχο ε, του ερυθρού τόνου. Ευχαρίστω να σα δώσω και άλλη διευκρινήση να απαντήσω σε ερωτήσει. Ευχαριστούμε. Και τώρα ο εισηγητή, όπω γνωρίζετε, είναι ο κύριο Ρωμέβα. Έχετε τον λόγο, κύριε Ρωμέβα. Ευχαριστώ. Εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλια της Επιτροπής επ' αυτού. Όπως γνωρίζετε σχεδιάζουμε να έχουμε και την, να παρακολουθήσουμε την επόμενη συνάντηση της ICAT που θα γίνει σε κάποιες εβδομάδες. Θα συζητηθούν εκεί κάποια πράγματα και βρισκόμαστε στην κατάσταση τώρα να πρέπει να ε, καλύψουμε αυτή την πτυχή. Υπάρχει μια τεχνική πτυχή που αφορά την ε, υλοποίηση της ε, συμφωνίας ε, από πλευράς ICAT όσον αφορά το πλαίσιο της ΕΕ, κάτι απόλυτα αναγκαίο να γίνει. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Από την άλλη πλευρά πάντα έχουμε σε σχέση με τα αλλιεύματα στοιχεία που χρειάζονται και θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό το πλαίσιο. Υπάρχει ένα περιθώριο ελιγμών που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση οποιασδήποτε απόφαση όπω αυτή. και το εκτιμώ ιδιαίτερα ότι έχει ανοιχτό πνεύμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη και θα πρέπει να αναμείνουμε να υπάρξουν κάποιες άλλες πτυχές μέχρι την υλοποίηση αυτής της συνεδρίασης να δούμε στο τέλος αν θα χρειαστούν κάποια θέματα που πρέπει να συζητηθούν για προσαρμογή κάποιων θεμάτων. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι σαφές και μπορούμε να κάνουμε αυτό το έργο σε τεχνικό επίπεδο αρκετά εύκολα και έτσι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στον κύριο Ρωμέβα να του πω ένα ανέκδοτο. Πριν από μερικές εβδομάδες ήμουν διακοπές στην Τουρκία και εμείς εδώ στην Επιτροπή μας πάντοτε μιλούσαμε για τη σημασία μικρομεσαίων στόλων αλλιευτικών και ακόμα και μέσα στο Πολδίπ ζητούσαμε από τους αλληλείς να χρησιμοποιούν τα μικρού μεγέθους αλλιευτικά πλοιάρια για τουρισμό. Ήμουν λοιπόν στο ΚΑΣ που είναι 1,5 χιλιόμετρο από το Καστελόριζο 1,5 χιλιόμετρο που θα μπορούσε κανείς να κολυμπήσει μέχρι εκεί. Αλλά στην τουρκική πλευρά έχουν εκατοντάδες μικρά πλοιάρια που πηγαίνουν τους τουρίστες βόλτα για να αλλιεύσουν τόνο. Και μίλησα με έναν τουρίστα που είπε ότι είχε πιάσει ένα-δύο τόνους και τους μαγείρεψε επιτόπου ο πλοίαρχος. Τι τόνο, bluefin μου είπε. Δύο τόνους φάγατε για το μεσημέρι, μα είπε ήταν μικρή. Εκατοντάδες πλοιάρια λοιπόν στις τουρκικές ακτές αλλιεύουν δεκάδες χιλιάδων κόκκινους τόνους και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Φαίνεται ότι ενώ ενθαρρύνουμε την μετατροπή της χρήσης των πλοιαρίων ε, αυτών για τον τουρισμό, από τη δική μας πλευρά πρέπει να σκεφτούμε και πώς θα μπορούσαμε να ελέγξουμε αυτή την αλεξέλεγκτη αλληλεία κόκκινου τόνου από εκτός κοινότητας. Ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε Στίβενσον. Η κυρία Πατράουν έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ ίδια θέλω να επιστήσω την προσοχή και να εκμεταλλευτούμε αυτή τη ευκαιρία για να απευθύνουμε, να ε, στοχεύσουμε την προσοχή σε μια πτυχή που θεωρώ πολύ σημαντική και συσχετίζεται με την ε, αλληλεία στις υπερ, ε, περιφερειακές περιοχές, στις απομονωμένες υπερπεριφερειακές περιοχές. Ε, σε σχέση με την αλληλεία του τόνου, αυτή γίνεται εκεί αποκλειστικά με την, ας με ένα πολύ επιλεκτικό τρόπο, ε, όσον αφορά τα είδη, όσον αφορά τα μεγέθη των αλλιευμάτων, την ποσότητά τους. Γι' αυτό όλοι γνωρίζουμε και είναι γνωστό ότι είναι φιλοπεριβαλλοντική αυτή η μέθοδος ε, βιο, ε, ε μικρής κλίμακας αλληλείας. Για τις υπερπεριφερειακές ε, περιοχές και τα στοιχεία που έχω εδώ είναι στη διάθεση ε, από πλευράς της δικής μου περιοχής των Αζωρών πρόκειται για πολύ μικρές ποσότητες που αλλιεύονται εκεί πράγματι και στον αλληλευτικό στόλο, τον ευρωπαϊκό αλληλευτικό στόλο, όταν έχουμε 7.500 τόνους, για παράδειγμα, η Πορτογαλία 225 ε, ε, όσον αφορά την, ε, τους τόνους αυτούς είναι ένα ελάχιστο ποσοστό. Τι συμβαίνει όμως αυτή τη στιγμή σε σχέση με αυτή την αλληλευτική δραστηριότητα. Συμβαίνει ότι τα στοιχεία όσον αφορά την περίοδο που διανοίγεται στις υπερπεριφερειακές περιοχές μας με ε, την ε, βιοτεχνική αυτή αλία ε, προβλέπονται σε σχέση με την 31η Οκτωβρίου όταν ε, έχει ήδη ε, εξαλειφθεί πλέον η δυνατότητα αυτού του αλλιεύματος και δεν υπάρχει αυτό το ψάρι εκεί. Ανοίγει λοιπόν αυτή η περίοδος αλλιεύσης όταν δεν υπάρχει τίποτα πλέον να αλλιευθεί εκεί. Και ποια είναι η επίπτωση για τους αλλιείς αυτής της κατάστασης. Οι κονσερβοποιητές, ε, η βιοτεχνία κονσερβοποίησης είναι υποχρεωμένη να αγοράζει τον τόνο από τα παραγαδιάρικα όταν έχει εκλείψει η δυνατότητα δική τους ε, ε, αλλιεύσει του δικού του, του, δικού τους είδους. Ε, δημιουργείται μια παράλογη κατάσταση. Οι ίδιοι οι αλείς των υπερπεριφερειακών περιοχών που έχουν πολύ μικρά σκάφη που επιλεκτικά με βιοτεχνική αλία αλλιεύουν σε ελάχιστες ποσότητες αυτό το είδος και δεν υπάρχει αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση από αυτές τις δραστηριότητες, τι κάνουν, δεν έχουν δυνατότητα να αλλιεύσουν αυτό το είδος και η δική τους ε, βιομηχανία υποχρεώνεται να αγοράσει το ψάρι αυτό για να το κονσερβοποιήσει από άλλους αλείς που δεν αλλιεύουν με βιοτεχνικό τρόπο και που αλλιεύουν ακριβώς τα ίδια ύδατα όπου οι ίδιοι οι ε, αλείς με, τη, τα βιοτεχνικά τους μέσα μικρής αλίας, παράκτειας αλίας αλλιεύουν. Είναι μια παράλογη κατάσταση διότι πραγματικά όταν περνάνε οι τόνοι από αυτά τα ε, ύδατα, από αυτά τα ε, χωρικά ύδατα οι ίδιοι δεν μπορούν να αλλιεύουν όμως τα παραγαδιάρικα από άλλες περιοχές μπορούν να τα αλλιεύουν. Βλέπουμε ότι εδώ ότι υπάρχει αρνητική επίπτωση για αυτούς τους αλείς. Ε, πρέπει να αγοράζουν το ψάρι σε ανώτερη τιμή από άλλους αλείς. Και εδώ βλέπουμε ότι επιβαρύνεται η βιοτεχνική αλληλεία λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Η μικρή κλίμακα αλληλεία και γι' αυτό θα δώσω και πιο εξειδικευμένα στοιχεία στον εισηγητή. Θέλω πραγματικά να ευαισθητοποιηθεί ο εισηγητής και οι παρόντες για μια κατάσταση που πραγματικά είναι παράλογη και άδικη. Και θα υποβάλω ας το πω έτσι, μια πρόταση τροπολογίας, τροποποίησης των στοιχείων, όχι αυξάνοντας την περίοδο, αλλά προσεγγίζοντας περισσότερο, ας το πω έτσι, το άνοιγμα της ε, διάρκειας της περίοδου για τους αλείς, ώστε να μπορούν εκείνοι να αλλιεύουν, οι επιτόπιοι αλείς, και όχι να αλλιεύουν οι εκτός περιοχής αλείς, και ε, να βρίσκονται οι γηγενείς σε αρνητική επίπτωση. Αυτό είναι το νόημα αυτής της ε, κίνησής μου να δούμε πώς μπορούμε, ας το πω έτσι, να υπάρξει ευαισθητοποίηση και κατονόηση από όλους για μια ειδική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος uh, is... Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι σαφές ότι υπάρχει το θέμα του πώς θα προστατεύσουμε τα είδη που αναφέραμε πολλές φορές εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε διαφορετικά είδη επιστημονικών δεδομένων. Άλλα μας λένε ότι αυξάνεται το απόθεμα, άλλα ότι κινδυνεύει. Επομένως στις δικές μας τουλάχιστον θάλασσες φαίνεται ότι δεν βελτιώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων. και πρέπει να ληφθούν μέτρα. Όπως είπε και ο κύριος Στίβενσον, το σημαντικό είναι πώς θα εφαρμοστούν επίσης. Και γι' αυτό η επόμενη συνάντηση θα μιλήσει ακριβώς για το θέμα του τρόπου εφαρμογής των μέτρων για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κάνουν, θα παίξουν το ρόλο τους όπως πρέπει γιατί πριν από μερικά χρόνια δεν συμφωνούσαμε ότι υπάρχει κίνδυνος για τα αποθέματα. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι μερικά ήδη βελτιώνονται τα αποθέματα τους, αλλά πρέπει να τα προσέξουμε όλα αυτά ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ κυρία Σένη. Κυρία Φράγα, θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι Κάνουμε λόγο εδώ για την υλοποίηση κοινοτικών προδιαγραφών μιας σύστασης, μιας τροποποίησης, ε, μιας σύστασης του ΙΚΑΤ όσον αφορά τον ερυθρόπτερο τόνο που το 2012 εγκρίθηκε και που μέσα σε ένα μήνα έχουμε και το θέμα της Ολομέλειας. Θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί, γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ στην κατάθεση αυτής της ε, πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεύτερο, θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα προβλήματα σε σχέση με την έκθεση των ε, αιτιολογικών σκέψεων, σε σχέση με τον καθορισμό των ΤΑΚ, που δεν έχει καμιά σχέση με τις ε, αλλιευτικές ε, περιόδους. Η Τουρκία όμως είχε αντίρρηση σε σχέση με το ΤΑΚ του ερυθρόπτερου τόνου και υπάρχουν και άλλα συμβαλόμενα μέρη τα οποία έχουν πρόβλημα με αυτό. Πώς λοιπόν είχε επίπτωση αυτό σε σχέση με τα ΤΑΚ του ερυθρόπτερου τόνου. Θέλω να ξέρω ποια είναι τα προβλήματα επίσης της και του καθορισμού ζωνών και περιφερειών. Ευχαριστώ. Εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Σύντομα. Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση ότι πραγματικά μας ε, έχουμε εδώ ένα θέμα, μια έκθεση, μια έκθεση που βρίσκεται και πρόθεσμα όσον αφορά τα, της αυτή τοποθέτηση. Τι θα κάνουμε, θα επικυρώσουμε μια και κάνουμε λόγο για, την, ε, για προηγούμενες περιόδους ε, που ολοκληρώνονται και σε σχέση με τα απειλούμενα ήδη και τα, το χρονοδιάγραμμα και τον καθορισμό ποσοστώσεων το θέμα είναι ότι είναι ένα πολύ περιπλοκό θέμα διότι όλα αυτά τα οποία μπορούν να ρυθμιστούν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των δικαιοδοσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ιδιαίτερα απαιτητικοί, σίγουρα. Όμως σε σχέση με άλλες χώρες ε, ή με άλλα κράτη που δεν αποτελούν ε, τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα. Προσυπογράφω απόλυτα την πρόθεση για ερώτηση της κυρίας Φράγκα. Αν υπάρχει μια χώρα όπως η Τουρκία που δεν συμφωνεί σε σχέση με την ποσόστοση θα συνεχίσει να αλλιεύει. Όχι μόνο γι' αυτό αλλά επειδή δεν, υπάρχει κανένα μέσο ελέγχου στο οποίο να υπάγεται. Το ίδιο γίνεται και με τους Κινέζους, τον στόλο των Κινέζων και τους Ταϊλανδούς, τους ε, Ταϊλανδέζους. Τι γίνεται εδώ σε σχέση με αυτές τις χώρες. Πρέπει να να υπάρχει μεγαλύτερος έλεγχος όσον αφορά τη μεταποιητική βιομηχανία, τις βιομηχανίες κονσερβοποίησης και για τα κεφαλόποδα είχε εκφραστεί παράπονο διότι ε, υπάρχει ε, περιορισμό σε σχέση με την ε, αλίευση στην ε, Μαυριτανία, αυξάνεται όμως ε, η δυνατότητα σε σχέση με την Κίνα και την Ταϊλάνδη. Να είμαστε συνεκτικοί στην προσπάθειά μας, να μπορούμε να λαμβάνουμε υπόψη για τα απειλούμενα ήδη τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη και το σύνολο, συνολικά την ευρύτερη εικόνα. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η προστασία των συμφερόντων μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα η Επιτροπή, παρακαλώ, θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που έγιναν. Thank you, Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ε, τα μέλη του Κοινοβουλίου για όλα αυτά που ρώτησαν και κυρίως να ευχαριστήσω τον κύριο Ρομέρα που είναι πολύ καλά ενημερωμένος για τον ερυθρό τόνο γιατί το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό στο παρελθόν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις Αζόρες και παρεμφερείς περιοχές. Στην ομιλία μου είπα ότι καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση στον ICAT μετά από μια επίπονη διαδικασία συζητήσεων. Βεβαίως ε, αυτό είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμού εσωτερικών συμβασμών, ε, συμβασμών με τα άλλα συμβαλόμενα μέρη. Αλλά ξέρετε, εμείς πιστεύουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα από τους ε, καλύτερους συμβασμούς που υπήρξαν για τον ερυθρό τόνο. Επίσης, είχαμε ε, πολλές συζητήσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, με τον κλάδο, με μικιό και πρόκειται να καταθέσουμε ένα περιεκτικό πακέτο. Πέρυσι το καταθέσαμε στον ICAT. Από τη μια ενισχύεται ο έλεγχος και από την άλλη υπάρχει η δυνατότητα οι στόλοι που αλλιεύουν ερυθρό τόνο να μπορούν να χρησιμοποιούν όσο μπορούν τις δυνατότητες που τους προσφέρονται για να διαπιστωθεί πώς μπορούν να μεγιστοποιηθούν οι ε, δυνατότητες. Δεν έχουμε ακούσει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα, ούτε πριν από τη συνάντηση της ICAT, για τις ε, συγκεκριμένες ε, περιοχές που θα ισχύουν σε αυτόνομες περιοχές σχετικά με τα ληφτικά εργαλεία. Και αυτό είναι κάτι που είχαμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν τα συζητήσαμε σε βάθος ε, με πολλούς και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Το δεύτερο που θέλω να απαντήσω έχει σχέση με το θέμα της ε, Τουρκίας, της αντιρρήσεις που υπάρχουν και επίση τις επιπτώσεις από αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Η Τουρκία διαφώνησε. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία διαφώνησε από τότε που έχουν συσταθεί τα ΤΑΚ και από τότε που υπάρχει το ε, πρόγραμμα αποκατάστασης του ερυθρού τόνου, το 2008 δηλαδή, μετά τροποποιήθηκε το 10 και το 12. Βέβαια, η Τουρκία ε, διαφώνησε μόνο για τα ΤΑΚ, όχι για τα άλλα θέματα που έχουν σχέση με τον έλεγχο και την παρακολούθηση κάποια άλλα στοιχεία του προγράμματος αποκατάστασης. Ε, εμείς ε, ως συμβαλόμενο μέρος, όχι ως Επιτροπή, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι όλα τα συμβαλόμενα μέρη της ε, Συμφωνίας Αλίας για τον Ερυθρό Τόνο ήδη το 2013 θα αρχίσουν να εφαρμόζουν τα νέα στοιχεία της αναπεριμένης απόφασης. Και αυτό επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του έτου σε μια συνάντηση του ICAT όπου ανεξάρτητα από την επίσημη θέση σε ισχύ της σύστασης που κατά κανόνα γίνεται έξι μήνες μετά τη λήψη απόφασης, δηλαδή τα συμβαλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι από την 1η Ιανουαρίου ε, θα εφαρμόζουν πλήρως τη σύσταση. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν η Τουρκία διαφώνησε, ε, δέχτηκε όμως η σύσταση να ισχύει και στην Τουρκία από την 1η Ιανουαρίου του 2013. Όπως σας είπα, αυτή είναι μια προαιρετική δήλωση και θα αναθεωρήσουμε την εφαρμογή του ελέγχου το 2013. Και κάτι άλλο, έχει σχέση με τα σχόλια σχετικά με τον τουρκικό έλεγχο και έλλειψη ελέγχου του στόλου αυτού. Ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για το πρόγραμμα αποκατάστασης του ερυθρού τόνου είναι ότι τα συμβαλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αποδίδουν και ένα κομμάτι της ποσόστοσής τους για την αλία αναψυχής. Βέβαια δύσκολο να το ελέγξει κανείς αυτό. Το 2012 η απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί πλήρως, ελήφθη και ενισχύσαμε και τον έλεγχο επιβάλλοντας τα συμβαλόμενα μέρη να διασφαλίσουν ότι η αλία αναψυχής αναπτύσσεται μόνο σε ένα κομμάτι του ΤΑΚ και με αυστηρά μέτρα. Ε, Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ε, θα δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Και θέλω να διαβεβαιώσω ε, τους ευρωβουλευτές ε, ότι εμείς δεν ενισχύουμε αυτή την αλή αναψυχής γιατί υπάρχουν προβλήματα με τον έλεγχο και όπως σας είπα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός αυτής. Θα συνεχίσουμε να τα ελέγχουμε και θα τα έχουμε κατά νου στη συνάντηση της Επιτροπής Συμβατότητας Compliance που θα λάβει η χώρα το Νοέμβρη. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω τον λόγο στον κύριο Ρομέβα για να ολοκληρώσει η συζήτηση επικεντρώνεται σε σχέση με τα υπεραπομονωμένα ε, περιφερειακά διαμερίσματα όπως είπε η κυρία Πατράων για τις Αζόρες ε, ε, για μας την Ισπανία για τις Κανάριες θα έχουμε στην πόλη του Ακροτηρίου στο Cape Town την συνάντηση, η επόμενη συνάντηση της ICAT που θα γίνει ε, για το 2013 και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και αυτές τις περιοχές όπως και τις ε, Κανάριες νήσους. Ο κύριος Ρωμέβα για να ολοκληρώσει τρία σχόλια σύντομα. Πρώτο, συμφωνώ γενικά και είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να τονιστεί στην επόμενη συνάντηση του ICAT πέρα από την ευρύτερη συζήτηση για τα τάξα που φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η επιστημονική σύσταση. Το μεγάλο πρόβλημα εξακολουθεί να είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος ε, και η εποπτεία αυτό αφορά και την Τουρκία φυσικά, αλλά επίσης και σε πολλές άλλες περιπτώσεις και σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Στόλο μεταξύ άλλων. Διότι αυτό που γίνεται υπάρχει συνεργασία για να την μπορέσουν να εκμεταλλευτούν κάποιες ζώνες. Υπάρχει ένα πρόβλημα λοιπόν εδώ σε σχέση με αυτό το θέμα και πρέπει σε σχέση με τις ζώνες της ΑΕΚΑΤ να εξεταστούν αυτά τα θέματα. Απαιτείται μια μεγαλύτερη δυνατότητα και κυρίως μεγαλύτερη πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα. Εξακολουθεί να είναι αυτό ένα κέριο θέμα. Δεύτερη πτυχή που θεωρώ την σημαντική και πρέπει να υπογραμμίσουμε την ανέφερε η κυρία Πατράων Νέβης. Είναι προφανές και επιμένουμε και μένουμε ότι οι επιπτώσεις ε, ε, κάποιων αλευτικών δραστηριοτήτων από πλευρά στόλων δεν είναι παντού οι ίδιες και υπάρχει μια πιο βιοτεχνική αλία, υπάρχει μια άλλη πιο βιομηχανική και γι' αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο να υπάρξουν συγκεκριμένοι περιορισμοί για κάποιε δραστηριότητε αλλιευτικέ που έχουν μεγαλύτερε επιπτώσει στα αλλιεύματα, όπω είναι η βιομηχανική αλία. Μέχρι σήμερα ισοπεδωτικά με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζαμε όλα τα ίδια αλληλείας ενώ δεν είναι ίδιας εμβέλειας και επίπτωσης όλες οι δραστηριότητες στην αλληλεία Πρέπει εδώ να διεξαχθεί λοιπόν μια συζήτηση. Είναι ακόμα ανοιχτά αυτά τα θέματα. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κλείσει η συζήτηση και πρέπει να δούμε τι επιπτώσει που υπάρχουν. Και τέλο ένα σημείο το οποίο δεν αναφέρθηκε προηγούμενα. Όμω ήθελα, θα ήθελα να το σημειώσουμε και αυτό. Αυτό αφορά τις διοργανικέ σχέσει ε, μεταξύ για παράδειγμα ημών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και έχουμε μια κάπω αξιοπερίεργη κατάσταση που δημιουργείται όταν εξετάζουμε την, σε σχέση με την εντολή ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξεταστεί και βλέπουμε σε σχέση με την επόμενη συνάντηση της ΆΙΚΑΤ από πλευράς της Επιτροπής απαιτείται να ακολουθηθούν μια ολόκληρη σειρά πρωτοκόλων με χεμήθεια και εμπιστευτικό χαρακτήρα ενώ ουσιαστικά η εντολή δεν ε, πρέπει να τροποποιεί ουσιαστικά εκείνα τα οποία έχουν συμφωνηθεί σε σχέση με μια δυναμική υπερβολική πρακτικών, ε, ας το πω έτσι, μέτρων ε, προστασίας κάποιων θεμάτων. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο πρέπει να εξετάσουμε και διμερώς να προετοιμάσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προετοιμάζοντας την επόμενη συνάντηση της ICAT στο Cape Town. Αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρωμέβα και σε σχέση με την ε, συνάντηση αυτή που χρειαζόμαστε για την προετοιμασία της ΑΕΚΑΤ συμμετέχουμε και πρέπει να γίνει αυτή η δουλειά από πλευράς του Κοινοβουλίου είμαστε απόλυτα στη διάθεση της Επιτροπής για να γίνει αυτό άλλος θέλει να παρέμβει όχι ολοκληρώθηκε η μερίσια διάταξη όσον αφορά τα θέματα της σημερινής πρωίας και στις 3 θα ακολουθήσει το επόμενο σημείο που απομένει. Ευχαριστώ λίγη συνεδρίασή μας.